Σήμασα για το θέμα της διάσκεψης των Παρισίων και ήρθατε στην Ολομέλεια. Σας καλωσορίζω θερμά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι, στις 12 Δεκεμβρίου πέρυσι στο Παρίσι είχαμε μια ιστορική ημέρα, ένα ιστορικό βήμα που επετεύχθη. Όλες οι χώρες της οικουμένης υποχρεώθηκαν να δώσουν την μάχη με δεσμευτικό τρόπο κατά της αλλαγής του κλίματος. Οι χώρες αυτές εκφράστηκαν με φιλόδοξους στόχους υπέρ του κλίματος. Η επιτυχία έχει πάντα πολλού πατέρε και γι' αυτό εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού, Κοινο... Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να ευχαριστήσω όλου εκείνου που επί πολλά έτη εργάστηκαν για την επιτυχία αυτή τη διασκέψεω τη Συνόδου των Παρισίων. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο κύριο Κανιέτε και την Λουξεμβουριανή Προεδρία και όλο το σύνολο δηλαδή τη ομάδα των διαπραγματευτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο εσεί κύριε Υπουργέ Λογόν Φαμπίου, είχατε μεγάλο μέρο σε αυτή την επιτυχία Καταφέρατε με τη διπλωματική δυνατότητα και ικανότητα που έχετε να συγκεράσετε τις διαφορετικές θέσεις. Καταδείξατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρόλο πρωτοπόρου και μπορεί να έχει ρόλο πρωτοπόρου για την προστασία του κλίματος και πρέπει να το κάνει αυτό. Τώρα είναι υποχρεωμένες οι χώρες αυτές τις δεσμευτικές υποχρεώσεις που ανέλαβαν να τις υλοποιήσουν, να επιτευχθεί δηλαδή η συμφωνία και κυρίως ε, είναι αδιαμφισβήτο ότι την υπόσχεσή μας ε, έναντι όλων πρέπει να τη στηρίσουμε. Η επιτυχία των Παρισίων δείχνει όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε πάρα πολλά να πετύχουμε. Γι' αυτό για μας είναι μεγάλη τιμή κύριε Υπουργέ ότι βρίσκεστε ανάμεσά μας. Αγαπητέ Λογάν Φαμπιούς, καλώς ήρθατε θερμά και έχετε τον λόγο αμέσως παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε Κανιέτε, Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, αγαπητοί φίλοι, καταρχήν θα ήθελα όλο ιδιαίτερω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Σούλς που με κάλεσε ω Πρόεδρο τη COP21 ώστε να σα παρουσιάσω τι βασικέ γραμμέ τη συμφωνία που υιοθετήθηκε στι 12 Δεκεμβρίου ε, του 2015 στο Παρίσι και να σας ε, ενημερώσω και για τα επόμενα βήματα. Το έτος 2015 ήταν δύσκολο σε ολόκληρο τον κόσμο και, και την Ευρώπη ε, ακόμη παρα, περισσότερο. Και γι' αυτό και η διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα αποτέλεσε μια ελπίδα. Επέτρεψε τη συγκέντρωση όλων των κρατών, των εθνών και έδειξε η διάσκεψη του Παρισιού ότι η διπλωματία και οι ε, πολυμερείς ε, διαπραγματεύσεις μπορούν να καταλήξουν σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Είχα δε έρθει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος για να σας και ότι θεωρούσαμε ότι θα ήταν μια καλή συμφωνία στο Παρίσι, αλλά τότε δεν γνωρίζαμε τα αποτελέσματα. Τώρα, διαμέσου των 29 άρθρων που περιλαμβάνει η Συμφωνία του, του Παρισιού και των 140 σημείων της απόφασης που τη συνοδεύει, αυτά τα κριτήρια για μια καλή συμφωνία πληρούνται. Καταφέραμε να έχουμε μια καθολική συμφωνία που βασίζεται σε εθνικές συμβολές 187 χωρών, η συμφωνία θεωρείται φιλόδοξη, συμπεριλαμβάνει μακροπρόθεσμα το περιορισμό της θέρμανσης του πλανήτη σε δύο βαθμούς, καθώς και τις προσπάθειες για τον περιορισμό σε 1,5 ε, βαθμό αλλά και την εξουδετερώση του άνθρακα μέχρι το τέλος του αιώνα. Ε, προβλέπεται ένας μηχανισμός πενταετούς αναθεώρησης των στόχων με πρώτο ραντεβού το 2023 αλλά έναν απολογισμό των προσπαθειών ήδη από το 2018. Πράγμα που θα επιτρέψει συζήτηση για να αυξηθούν οι δεσμεύσεις σε σχέση με τη συνέχεια που θα δοθεί στις δεσμεύσεις. Ένα κοινό πλαίσιο διαφάνειας έχει καθοριστεί με αυτό που ονομάζουμε ευελιξία ανάλογα με τις ικανότητες κάθε χώρας τις δυνατότητες κάθε χώρας. Η συμφωνία είναι δεσμευτικός, ε, νομικός δεσμευτική όσο μπορούμε να πετύχουμε δεσμευτικές ε, πολιτικές από διάφορα κράτη και η συμφωνία εν γέννη αναγνωρίζεται ως δίκαια. Η έννοια της διαφοροποίησης ε, διαπνέει όλα τα θέματα και η αλληλεγγύη των πλούσιων χωρών θα λειτουργήσει προς τις πιο ευάλωτες χώρες με δέσμευση να σεβαστούμε και να ξεπεράσουμε τον στόχο των 100 δις δολαρίων ετησίως υπέρ των ευάλωτων χωρών και να οριστούν πριν από το 2025 συγκεκριμένα όρια. Τα αποτελέσματα αυτά τα οποία πολύ λίγος κόσμος πίστευε ότι θα επιτευχθούν πριν από την COP21, οφείλει πολλά στου Ευρωπαίους. Όπως το είπατε και εσεί, κύριε Πρόεδρε Σούλτ, ε, ιδιαίτερα το επίπεδο φιλοδοξίας της συμφωνίας ε, και θα ήθελα να χαιρετήσω την δέσμευση που ε, περιλαμβανόταν στην έκθεση του κυρίου Μπαρνιό, που είναι εδώ παρόν, που έχει τίτλο «Προς μια διεθνή συμφωνία στο Παρίσι», την οποία υιοθετήσατε την έκθεση αυτή τον Οκτώβριο του 2015, πριν τη διάσκεψη δηλαδή, και επίσης την ισχυρή δέσμευση του Επιτρόπου Καλνιέτε, με τον οποίο θα σας πω ότι ε, περάσαμε πολλές λευκές νύχτες ε, και να ευχαριστήσω και την ε, Προεδρία του Λουξεμβούργου, την Υπουργό Καρόλ Γεσμούρ που μας, ε, που βοήθησε πάρα πολύ, αλλά και κάθε μια από τις χώρες σας που επέτρεψε να φτάσουμε σε αυτή την επιτυχία. Η COP21 επέτρεψε να συνδεθούν με τα κλιματικά ζητήματα για πρώτη φορά σε αυτή την κλίμακα ένα σημαντικό αριθμό μη κυβερνητικών φορέων. Πάνω από 5.000 πόλεις, περιφέρειες, επιχειρήσεις, επενδυτές και ΜΚΟ που προέρχονταν από 180 χώρες ανέλαβαν δεσμεύσεις με αυτή την ευκαιρία. Δηλαδή υπάρχει η κρατική πτυχή και η μη κρατική πτυχή πολλά φιλόδοξα προγράμματα, των οποίων αντίκτυπος θα πρέπει να καταμετρηθεί πριν από το 2020 και ξεκίνησαν πριν από την διάσκεψη στο σύνολο. Πιστεύω πως μια δυναμική μετακίνηση ξεκίνησε προς την ε, ανάπτυξη χωρίς άνθρακα. Αυτός ο μηχανισμός ε, είναι αναπόδραστος, ιστορική σημασία λέμε συχνά, αλλά πιστεύω πως και πάλι αυτός ο όρος εδώ δεν είναι ο καταλληλότερος και ότι στον απαραίτητο ε, αγώνα κατά της ε, κλιματικής απορρίθμισης θα υπάρχει το πριν το Παρίσι και μετά το Παρίσι. Βέβαια πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα ώστε να διευκρινιστούν και να, ε, να διευκρινιστεί και να εφαρμοστεί αυτή η ιστορική σημασία σε συμφωνία. Το 2015 ήταν η χρονιά των διαπραγματεύσεων και των αποφάσεων και το 2016 θα πρέπει να είναι η χρονιά των τεσσάρων ε, στόχων, δηλαδή διαδικασία υπογραφής και κύρωσης. 22 Απριλίου στον ΟΗΕ θα αρχίσει θα ανοίξει μάλλον η συμφωνία για ε, ε, ε, συνυπογραφή. Οι χώρες που αντιπροσωπεύουν το 55% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να την υπογράψουν για να μπορέσει να αρχίσει να ισχύει αυτή η συμφωνία. Και θα πρέπει βέβαια και ένας μεγάλος αριθμός, όσο γίνεται μεγαλύτερος, από τις ευρωπαϊκές χώρες να είναι παρόν Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να δίνει το παράδειγμα υπογράφοντας τη Συμφωνία του Παρισιού από τις 22 Απριλίου και έπειτα κυρώνοντας την ίδια συμφωνία όσο γίνεται πιο σύντομα. Δεύτερο στόχο είναι οι διευκρινήσει όσον αφορά τη Συμφωνία του Παρισιού αλλά και την απόφαση που την συνοδεύει. Το Δεκέμβριο ετέθηκαν οι αρχέ και οι συγκεκριμένοι στόχοι. Τώρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τον τρόπο υλοποίησή του. Αυτό θα είναι το αντικείμενο της πρώτης συνεδρίασης της ομάδας που θα προετοιμάσει τις εφαρμοστικέ αποφάσεις στην Βόνη τον Μάιο, ώστε να έχουμε συγκεκριμένες ε, ε, διαδικασίες για τη χρηματοδότηση αλλά και για την ε, πενταετή αναθεώρηση των εθνικών δεσμεύσεων αλλά θα πρέπει να ορίσουμε και κανόνες για τη διαφάνεια στη παρακολούθηση και στην υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων ο στόχος ε, παραπέμπει στην περίοδο πριν το 2020. Πέρα από την εφαρμογή της συμφωνίας, τη οποία η έναρξη ισχύω προβλέπεται το 2020, θα χρειάζεται μια διαδικασία σε σχέση με τις δράσεις που θα πρέπει να γίνουν πριν από το 2020. σχεδιο δράση δράσης Λίμα-Παρίσι που περιλαμβάνει και του μη κυβερνητικού φορεί. Α πούμε, διεθνή ε, Ηλιακή Συμμαχία που ξεκίνησε από τον ε, Ινδό Πρωθυπουργό και ε, όπου συγκεντρώνει σχεδόν όλες τις χώρες ανάμεσα στο τροπικό του εγώκερου και το τροπικό του καρκίνου. Έπειτα, άλλοι επενδυτές ε, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για την ανάπτυξη των καθαρών τεχνολογιών, μεταξύ των οποίων και ο Bill Gates. Επίσης, ε, ε, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίηση απέναντι στις καταστροφές, το σύστημα COOLS όπω λέγεται, και το σύστημα κλιματική εξασφάλισης για τις ευάλωτε χώρε, επί το οποίο έχει εργαστεί πολύ η Γερμανία. Προστασία δε των τροπικών δασών και θέλω να επιμείνω για τι οικονομικές μας δεσμεύσεις απέναντι στι ανανεώσιμες πηγέ ενέργεια στην Αφρική που θα πρέπει να ανανεωθούν σύντομα. Για όλες αυτές τις δεσμεύσεις θα πρέπει λοιπόν να γίνουν πρόοδοι ήδη από φέτος. Τελευταίο στόχο είναι η προετοιμασία τη COP22 που θα γίνει στο Μαρακέ στα τέλη του 2016 και θα συνεργαστούμε με του μαροκινού φίλου μα στο ίδιο πνεύμα όπω οι Περουβιανοί είχαν συνεργαστεί μαζί μα για να προετοιμάσουμε το COP21 και έτσι να έχουμε και εκεί επιτυχία στο Μαρακέ τον Νοέμβριο μαζί με τους μαροκινούς φίλους και ένα σωρό ε, διεθνών ηθινόντων θα κάνουμε άτυπες και επίσημες ε, συσκέψεις για την ε, μέθοδο ε, που θα μας οδηγεί στην επόμενη στη διάσκεψη. Πέρα από αυτούς τους τέσσερις στόχους θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε σημαντικούς τομείς που δεν καλύπτονταν από τη Συμφωνία του Παρισιού αλλά στους οποίους πρέπει να υπάρξει δράση. Αεροπορικές μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές και μια συμφωνία επί της αρχής που εν μέρη είχε γίνει με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ που στόχο έχει να περιορίσει το αέριο FFC που συμβάλλει στη δημιουργία του θερμοκηπίου. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είναι εύκολο, αλλά η επιτυχία του Παρισιού και ο επίγοντα χαρακτήρα ε, των απαραίτητων δράσεων θα πρέπει να μα επιτρέψουν να επιτύχουμε αποτελέσματα. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, στην πολλά υποσχόμενη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά από το Παρίσι, είμαι πεπισμένο και ελπίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει τη δέσμευσή τη στην υπηρεσία τη ε, ε, διατήρηση του πλανήτη μα. Ω προ αυτό, νομίζω θα πρέπει να αναλυφθούν πολλέ πρωτοβουλίε. Η πρώτη αφορά την κύρωση από πλευρά Ένωση τη τροπολογία τη Ντόχα που σχετίζεται με τις δεσμεύσεις για τη δεύτερη περίοδο του πρωτοκόλλου του Κιώτου. Υπάρχουν μόνο λίγε χώρε που δεν έχουν ακόμα κυρώσει ε, και θα πρέπει να το πράξουν σύντομα. Άλλη πρωτοβουλία που θα πρέπει να αναλυφθεί από την Ένωση, τις δεσμεύσεις για το 2030. Μας περιμένουν διάφορες διαπραγματεύσεις, ας πούμε η μεταρρύθμιση της αγοράς εκπομπών άνθρακα, το ETS, αλλά και ε, σε τομείς που δεν εξαρτάται από το σύστημα ETS, όπως οι μεταφορές ε, ή οι οικοδομές. Για την πρώτη αδέα ανάγνωση της αναθεώρησης της οδηγίας ETS θα πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ενέργεια για να προωθηθεί ενεργειακή μετάβαση στην ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιμένοντας και στις νέες θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν, γιατί αυτό τα όλα δεν είναι μόνο μια δέσμευση, είναι και μια μεγάλη ευκαιρία. Διάφορα κείμενα θα κατατεθούν από την Κομισιόν μέσα στο 2016 ώστε να προχωρήσει αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα. Α πούμε, ενίσχυση των δεσμεύσεών μα σε σχέση με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ή την ενεργειακή απόδοση και αποτελεσματικότητα. Και εδώ βασίζομαι στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προχωρήσουμε γρήγορα. Τέλος, θα πρέπει να ε, θαρρύνουμε ε, την βιώσιμη ανάπτυξη στους νότιους εταίρους μας. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να, ε, να προωθήσει και να στηρίξει τις χώρες αυτές οικονομικά, τεχνολογικά, αλλά και με την εμπειρογνωμοσύνη της. Η διάσκεψη του Παρισιού είναι λοιπόν αναμφίβολα μια επιτυχία στον αγώνα κατά της κλιματικής απορρίθμισης, ακόμα και αν δεν είναι η καταληκτική ημερομηνία. Οι δράσεις θα πρέπει να συνεχιστούν και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, φέρει μεγάλη ευθύνη στις μελλοντικέ εργασίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο ώστε να ε, προωθήσει όλες τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα υπογραμμίσω κάτι το οποίο δεν θυμίζουμε συχνά, αλλά το οποίο θεωρώ σημαντικό. Η Συμφωνία του Παρουσιού δεν αφορά μόνο το κλίμα με τη στενή του αέρια, αλλά το ε, γενικό περιβάλλον, την βιοασφάλεια, ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αλλά επίσης είναι και μια συμφωνία υπέρ της ασφάλειας και της ειρήνης. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ η ε, έλλειψη τροφίμων και νερού, οι μαζικές μετακινήσεις λόγω των κλιματικών αλλαγών, οι απειλές ε, λόγω των ρηκτών καυσίμων, ε, ανεξέλεγκτη απορρίθμιση του κλίματος θα οδηγούσε σε γενικευμένες σειράξεις. Αρνούμενοι όπως το κάναμε και στο Παρίσι, αυτή την κατάσταση και ανανεώνοντας τη δέσμευσή μας για τις υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις απαλλαγές από τον άνθρακα, θέλουμε να λειτουργήσουμε ως ε, ε, ένα κέντρο ειρήνης ε, έναντι μιας χαοτικής και αβέβαιης απορρίθμισης του κλίματος. Για μας κάτι τέτοιο είναι σημαντική συνιστόσα της συμφωνίας του Παρισιού που η Ευρώπη έπαιξε και θα συνεχίσει να παίζει πλήρως το ρόλο της. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε θερμά κύριε Υπουργέ. Τώρα θα λάβει τον λόγο εξ ονόματος του ΕΛΚ ο κύριος Λίζε παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα και εγώ πρώτα πρώτα στον κύριο, τον κύριο ε, Φαμπιού να τον ε, συγχαρώ θερμά. Ο τρόπος με τον οποίο ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων ήταν ένα από τα κλειδιά που οδήγησαν σε μια επιτυχή συμφωνία των Παρισίων. Πολύ καλά δράσατε και όλη την ενέργεια και το πολιτικό σας βάρος το ρίξατε στην πλάστιγκα για να το πετύχετε αυτό. Αλλά ευχαριστώ επίσης και προσωπικά, Πρόεδρε, και τις, για τις ευχαριστίες ε, προς τον κύριο Επίτροπο Μιγέλα Ριασκανιέτε και από πλευρά ε, του συναδέλφου των ε, Πρασίνων ε, όταν ήρθε η ώρα επένου κατά το παρελθόν στον κύριο Κανιέτε. Θυμάμαι τις αντιπαραθέσεις που υπήρχαν ο κύριος Επίτροπος ε, έκανε καλή δουλειά και πριν από το Παρίσι και στο Παρίσι έκανε εξαιρετική δουλειά και πέτυχε το στόχο. Και συμφωνώ μαζί σας κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, έχει σπουδαιότητα αυτή η συμφωνία, όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αυτά τα δύσκολα χρόνια που ο κόσμος ανησυχεί και βρίσκεται σε ταραχή ότι τα καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία όπου εν μέρη χώρες υποχρεώθηκαν, δεσμεύθηκαν από κοινού ακόμα και παρόλες αντιπαραθέσεις και τριβές να συμφωνήσουν σε ένα κοινό στόχο. 195 χώρες συμφώνησαν για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα την ανακούφιση της ατμόσφαιρας και είναι σημαντικό Έχω κάποιες ε, ωστόσο επιφυλάξεις όσον αφορά τον στόχο της αναχέτησης της θέρμανσης του πλανήτη στο, σε 1,5 ε, βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να πούμε ότι <clears throat> δεν υπάρχουν αρκετές δεσμεύσεις, ε, δεν υπήρχαν αρκετές δεσμεύσεις για 2% και θα θέλαμε το 2 το, το, οι δύο βαθμοί υπερθέρμανσης να επιτευχθούν ώστε να έχουμε προοπτικές για το μέλλον και αναφερθήκατε στο θέμα των μεταφορών και των ναυτιλιακών μεταφορών που και αυτές πρέπει να ε, εμπλέκονται και να ρυθμίζονται όσον αφορά τις εκπομπές τρύπων τους και πρέπει να δοθεί στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό αυτή η εντολή. Κρίμα που δεν το καταφέραμε αλλά χαίρομαι για το ότι αναφέρατε ότι πρέπει να γίνει κάτι για αυτούς τους τομείς και θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά με την κυβέρνησή σας επίσης όπως ε, και για την Γερμανία που γνωρίζω καλύτερα να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε νομοθετικό έργο στην Ευρώπη. Και όταν ε, η διεθνή ε, Οργάνωση Αεροπορικών Μεταφορών ICAO δεν είναι σε θέση να πετύχει μια μείωση των εκπομπών ρήπων του θερμοκηπίου, μείωση και όχι σταθεροποίηση, ε, τότε πάλι θα έχουμε πρόβλημα και δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε αξιόπιστοι. Δεν είναι δυνατόν όλοι να καταβάλουν προσπάθειες με ιδιαίτερη δραστηριότητα και προσπάθεια για να τα καταφέρουμε με φιλόδοξους στόχους και άλλοι τομείς να διαφορούν και να μην καλύπτονται. Εδώ πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να είμαστε δίκαιοι στις φιλοδοξίες μας και στον επιμερισμό του έργου ώστε οι στόχοι μας να μπορέσουν να επιτευχθούν χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση από ε, κάποιους μόνο. Έχουμε λοιπόν πολύ σκληρή δουλειά μπροστά μας. Σας ευχαριστώ για όλα. Σας ευχαριστούμε κύριε Λίζε. Για τους σοσιαλδημοκράτες θα λάβει τον λόγο η κυρία Φανμπρέμπτ παρακαλώ. Κύριε Φαμπιούς, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοινοβούλιο. Καταρχάς, δεν είναι πρωτότυπο αυτό, αλλά θέλω να σας συγχαρώ εν ονόματι όλης της ομάδας για την έξοχη δουλειά που επιτελέσατε σαν Γαλλική Προεδρία. Ο τρόπος που προετοιμάσατε την ΚΟΠ, το πώς την χειριστήκατε, ήταν ένας λαμπρός, εξαιρετικός ε, και πετύχατε αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε διότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπαιξε σημαντικότατο ρόλο, κατάφερε να διατηρήσει ψηλά τις φιλοδοξίες, δημιουργήσατε γέφυρες προς τις ε, διάφορες συμμαχίες στις διαπραγματεύσεις και υποστηρίξατε την Γαλλική Προεδρία και ίσως ο συνδυασμός των δυο σας ε, οδήγησε στην επιτυχία. Αυτό δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί, είναι σημαντικότατο. Για πρώτη φορά στο Παρίσι σχεδόν όλες οι χώρες, σε όλο τον κόσμο, αναπτυσσόμενες χώρες και αναδυόμενες οικονομίες δεσμεύτηκαν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Εν αυτή τη ενία το Παρίσι είναι η πρώτη παγκοσμίω βελία συμφωνία και αυτό είναι κρισίμου σημασίας για το μέλλον. Αναφερθήκατε και εσείς αυτό. Λοιπόν, ότι τελικά το 2015 ήταν μια φρικτή χρονιά. Τα προβλήματα στη Μεσανατολή Πόλεμη, η Ουκρανία, η κρίση των προσφύγων και επιθέσεις στο Παρίσι. Ήταν άνω Και φάνηκε διχασμένος, διρεμένος ο κόσμος και η Ευρώπη. Η συμφωνία του κλίματος ε, άλλαξε το κλίμα που επικρατούσε και δημιουργεί κάποια συνδοξία για το μέλλον. Και η πόλη του φωτός, το Παρίσι, έγινε η πόλη της ελπίδας και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Όμως δεν ήταν τα πάντα επιτυχή, πρέπει να το παραδεχτούμε. Ένα παράδειγμα χτυπητό είναι η διεθνή τομέα της αερομεταφορών και της ναυτιλίας. Πολλές εκπομπές προέρχονται αυτούς τους δύο τομείς και συγκρίνονται αυτές οι εκπομπές με τις εκπομπές της Νοτιού Κορέας και της Γερμανίας μαζί. Και αυξάνονται αυτές οι εκπομπές αερομεταφορών και ναυτιλίας. Το επόμενο έτος θα αυξηθούν οι εκπομπές κατά 2.070% και πρέπει να πούμε ότι αποτύχαμε που δεν συμπεριλάβαμε τους τομείς αυτούς στη συμφωνία. Η ερώτησή μου προς εσάς και στους δύο, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό τον επόμενο χρόνο. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι δύο σημαντικότατοι τομείς θα συμμετάσχουν και αυτοί σε μελλοντική εφαρμογή των μέτρων. Δεν συμφωνώ με τον συνάδελφο του ΕΛΚ Πιστεύω ότι η συμφωνία για τους δύο βαθμούς και η προσπάθεια για τον 1,5 βαθμό είναι σημαντικότατη. Αν θέλουμε μπορούμε να πετύχουμε το στόχο. Αλλά αυτό θα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε ότι την Ευρώπη. Έχουμε μια καλή συμφωνία επί χάρτου όμως. Αν θέλουμε να πετύχουμε θα πρέπει να την εφαρμόσουμε. Άρα αυτό σημαίνει, και στέφω προς τον Επίτροπο, μεγαλύτερες φιλοδοξίες, καλύτερους, πιο φιλόδοξους στόχους από ό,τι μέχρι τώρα. Είχαμε στόχους για το 2030 και το 2050. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι πήραμε τη χαμηλότερη συνιστόσα των στόχων όταν έγιναν υπολογισμοί τα IPCC. Είπαμε 2050 80%. Να πάμε σε υψηλότερους στόχους και να εξασφαλίσουμε το ότι οι εκπομπές μας θα μειωθούν κατά 95% μέχρι το 2050. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, αλλά μπορούμε να κοιτάξουμε προς τον κόσμο μόνο αν επομιστούμε τις δικές μας ευθύνες. Τα απευθύνω αυτό και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πότε θα δούμε περαιτέρω εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει αυτά να γίνουν πριν ολοκληρωθεί η αναθεώρηση της ισχύουσης νομοθεσίας όπως αναφέρθηκε το ETS. Κλείνοντας, στρέφομαι προς εσάς, κύριε Φαμπιούς, εκ νέου, για να προβώ στο τελικό μου σχόλιο. Σας είμαι για το επιτελεστέν έργο. Όπως πανέφερα, έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Δεν είστε μόνο πρόεδρος της COP21, αλλά και υπουργό εξωτερικών σημαντικότητα του κράτους μέλους έχετε ηθική ευθύνη μαζί όλους μας. Υπέχετε ηθική ευθύνη να υπομειστείτε την ευθύνη σας. Και βασιζόμαστε πάνω σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Φανμπρέμπτ. Για τους Ευρωπαϊκούς Συντηρητικούς ο κύριος Ντάνκαν τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ υπέροχο, έξοχο αποτέλεσμα αυτό των Παρισίων. Έχω την εντύπωση ότι μετά, αντί να γιορτάζουμε και να επαναβογόμαστε στις δάφνες μας, πολλοί άρχισαν να σκέφτονται τι είχαν συμφωνήσει την προηγούμενη νύχτα. Διότι στην πραγματικότητα κάποιες συμφωνίες είναι αρκετά εξαιρετικές. Είναι σαν να ψάχνει κανεί να βρει κανεί τα περίεργα SMS ή τα tweet που έστειλε κανεί στο τηλέφωνό του. Έτσι και εμεί ανακαλύψαμε ότι εδώ τη τολμηρή αυτή συμφωνία εμπεριέχεται πραγματική τολμηρότητα. Αυτό το όριο του 1,5, το 1,5 βαθμού που αναφέρθηκε. Άκουσα ένα συνάδελφο μιλάει υπέρ και έναν κατά. Ό,τι και να συμβαίνει, προχωρούμε με κάποιο ρυθμό. Πρέπει να έχουμε υπόψη τον προορισμό προ τον οποίο κινούμεθα. Οι φιλοδοξίε Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής αντιπροσωπεύουν μόλι το 70% τη προσπαθία επίτευξη των στόχων του 2020. Και αυτή η φιλοδοξία πρέπει να επανεξεταστεί. Απευθύνομαι προ τον Επίτροπο τον κύριο Κανιέτη. Πρέπει να ευχαριστούμε για τα αποτέλεσμα στο Παρίσι. Δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον τον άνθρακα, σύμφωνα με τη συμφωνία. Πολύ σοβαρέ προκλήσει για το Κοινοβούλιο. Πρέπει να στερνιστούμε τι προκλήσει και να ανταποκριθούμε στι προκλήσει των Παρισίων. Συγχαρητήρια. Έκτακτο το επίτευγμα σα στο Παρίσι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντάνκαν. Για τους φιλελεύθερους τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριος Γερμπράντη παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Υπουργό τον κύριο Φαμπιούς έξοχος ο ρόλος που διαδραμάτισε στο Παρίσι στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία. Πραγματικά είναι μια ιστορική συμφωνία. Έστειλε σαφές μήνυμα. Δείχνει ότι ο κόσμος αμετάκλητα κινείται προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Συμφωνώ με εκείνους που λέγουν ότι το Παρίσι είναι απλώς μια συμφωνία πιχάρτου. Όμως δεν να μην λησμονούμε και την αξία του χαρτιού. Χρειαζόμαστε το χαρτί, τη συμφωνία πιχάρτου, για να κινηθούμε πραγματικά επιτόπου να δραστηριοποιηθούμε. Αναφερόμενο σε δράση, όπως και Πέτερ Λίζε και εγώ, θα ήθελα να τονίσω κάτι. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα από αυτά που συμφωνήσαμε στο Παρίσι όχι μόνο για να μείνουμε κάτω από το όριο των δύο βαθμών, αλλά και πιο σημαντικό να πλησιάσουμε το στόχο του 1,5 βαθμού. Μιλώντα για δράσει, θέλω να επικεντρωθώ επί των δράσεων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Έχουμε τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Αρκούν όμω εν συγκρίση με τη Συμφωνία των Παρισίων. Τι γίνεται με τη διαρροή άνθρακο. Η ιδέα τη διαρροή άνθρακο βασίζεται στην εξή υπόθεση. Ότι ο υπόλοιπο κόσμο δεν κάνει αυτά που κάνουμε εμεί. Αυτό θα αλλάξει τώρα. Τι θα κάνουμε λοιπόν για τη διαρροή άνθρακα, τι γίνεται για τους στόχους 2020, 2030, 2050, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε βάλει ένα όριο 1,5 βαθμού. Προσβλέπω στα σχόλια του Υπουργού του κ. Φαμπιούς. Πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσει τις προσπάθειές της. Τέλος κύριε Πρόεδρε, θέλω να μιλήσω για την ανταγωνιστικότητα. Η Συμφωνία των Παρισίων ξεκαθάρισε κάτι όσον αφορά την οικονομία μας. Τι, ότι η χαμηλή κατανάλωση του άνθρακα θα είναι κάτι πιο ανταγωνιστικό από την υψηλή κατανάλωση άνθρακα. Αυτό είναι πολύ σημαντική, κρίσιμη έννοια. Παράδειγμα, ιστορική στιγμή αυτή την εβδομάδα είχαμε στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ μια εταιρεία που ηγείται στη βιωσιμότητα, η Unilever, για πρώτη φορά στην ιστορία, έγινε, αυξήθηκε σε αξία από μια εταιρεία που δεν θεωρείται ότι ηγείται στην προσπάθεια, την Royal Dutch Shell. Ιστορική στιγμή και δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση. Μιλώντας για ανταγωνιστικότητα, έχω κάποια ανησυχία. Κύριε Υπουργέ, κύριε Φαμπίους, γιατί η Ευρώπη αρχίζει να υστερεί όσον αφορά τις επενδύσεις σε καθαρή τεχνολογία. Ερώτησή μου, πιστεύετε για να διαφυλάξουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειες προς μια οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γεμπράντη. Για την ενωτική αριστερά, η κυρία Μινέρ, παρακαλώ. Yes, thank you. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Φαμπιούς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι ήρθατε εδώ στο Στρασβούργο. Δεν μπόρεσα να σας συγχαρώ πριν, αλλά τα αποτελέσματα από το Παρίσι, από το Δεκέμβριο είναι κάτι για το οποίο θα σας ευχαριστήσω εδώ. Γνωρίζετε τι έλεγε Μπίλι Χόλιντε, το δύσκολο το κάνουμε τώρα και στο μέλλον ίσως όμως πετύχουμε τα ανέφικτο. Αυτό έλεγε Billy Holiday. Κάναμε το πιο δύσκολο και θα πρέπει να πετύχουμε τα ανέφικτο τώρα. Πολλά απομένουν να κάνουμε. Η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη. Πρέπει να απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα, να κινηθεί προς εναλλακτική βιώσιμη ενέργεια, ενεργειακές πηγές βιώσιμες. Πρέπει να εργαστούμε καλύτερα όσον αφορά τη χρήση των ενεργειακών πόρων. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις κατοικίες. Η χαμηλή τιμή του πετρελαίου είναι ένας καλός τρόπος για να απαλλαγούμε από τις επιδοτήσεις που χορηγούνται στα ορυκτά καύσιμα. Όλα αυτά μπορώ να τα υποστηρίξω. Ας είμαι θα όμως ειλικρινής. Από πλευρά Ολλανδική Προεδρία δεν περιμένουμε πολλά. Την περασμένη εβδομάδα μίλησα με την κυρία Σάρον Ντέξ, την Υπουργό, την Αρμόδια και τη ρώτησα τι θα κάνουμε μετά το Παρίσι. Αύριο μάλλον σήμερα το πρωί, μιλήσαμε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μαρκ Ρούτερ, και είδαμε ότι δεν είναι κατά της εισαγωγής της τεχνολογικής πρόοδου. Χρειαζόμαστε όμως κάποιον να ηγηθεί. Πρέπει να ηγηθεί η Ευρώπη. Ριζοσπαστική ηγεσία απαιτείται για να πετύχουμε βιώσιμα αποτελέσματα. Η προεδρία σας της ΚΟΠ θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους ε, στο Μαρακές και ζητώ από εσά, αν μπορείτε, να βοηθήσετε να πετύχουμε το ανέφικτο. Το αδύνατο. Το 2015 έγιναν διαπραγματεύσεις, πετύχαμε αποτελέσματα. Το 2016 θα είναι το έτος της εφαρμογής, της υλοποίησης, της δράσης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, στη σωστή κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι η Ευρώπη και η Ολλανδική Προεδρία θα συνεχίσουν με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε. Τον λόγο θα λάβει τον λόγο εξ των Πρασίνων ο κύριος Ζαντό. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ θα έπρεπε να ήσασταν εδώ ω προσκεκλημένο, νομίζω, στη διάρκεια της ψηφοφορία, όταν το σύνολο των Ευρωβουλευτών είναι παρόντες ε, και τόσο που είναι σημαντικό αυτό το θέμα, που αξίζει να συζητείτε ενώπιον όλων των Ευρωβουλευτών. Όλοι σας συνεχάρισαν και δικαίως εσά και την ομάδα σας για την πολύ καλή δουλειά που έγινε στο Παρίσι. Και ελπίζω πω θα μπορέσετε να μεταβιβάσετε στον επόμενο Πρόεδρο την ποιότητα της εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκατε, γιατί πιστεύω πως επίσης επανεφίβρατε ε, μια μορφή προεδρίας της ΚΟΠ. Συχνά λέγεται ότι στην αρχή διστάσατε όταν έπρεπε η Γαλλία να υποβάλει την υποψηφιότητά της. Είμαι απόλυτα πεπισμένο σήμερα πως ζήσατε ε, κάποιες από τις πιο έντονες στιγμές της σταδιοδρομίας σας. Ε, προφανώς η COP21 με το στόχο της να προσεγγίσει τον 1,5 βαθμό σας επιβάλλει να βγείτε, να απομακρυνθείτε από τις ορυκτές ενέργειες. Ε, αυτή η συμφωνία είναι αδύναμης δέσμευσης. Θα δούμε πώς θα οικοδομηθούν οι εφαρμοστικές διατάξεις. Οπότε βασικά εδράζεται σε τους κύκλους που θα μας μετακινήσουν από το 3, βαθμού σήμερα που είναι το κλιματικό χάος προς το 1,5 βαθμό. Αλλά για να λειτουργήσει ένα τέτοιο ε, ενάρετο κύκλο θα πρέπει όλοι να βάλουν τα δυνατά τη. Οι προποθέσει είναι ε, πιο ευνοϊκέ από ό,τι ποτέ. Σήμερα βλέπουμε σε ποιο βαθμό οι ανανεώσιμε ε, πηγέ ενέργεια όπω η φωτοβολταϊκή, η ολική είναι οι πιο θετικέ ενώ το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο η πυρηνική ενέργεια και σύντομα και ο άνθρακας. Όμως όταν βλέπουμε τα τελευταία νούμερα για τις επενδύσεις ε, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βλέπουμε πως όλες οι περιφέρειες του κόσμου προχωρούν στις επενδύσεις τους εκτός από την Ευρώπη και κυρίως λόγω της Γαλλίας, όπου οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά το ίμιση το 2015, τη στιγμή όπου αναπτύσσεται παντού αλλού. Και επί τότε ακούσαμε τη σημερινή συζήτηση το πρωί, στην παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας, μια φράση μόνο υπόθηκε για το κλίμα, μόνο μια φράση για το κλίμα. Αν αυτή είναι η ατμόσφαιρα στο Συμβούλιο για το κλιματικό ζήτημα, φοβούμε πως τελικά αυτός ο ενάρτητος κύκλος ανάμεσα στα κράτη, τις επιχειρήσεις, ε, τις ε, περιφερειακές ε, οργανώσεις κτλ. δεν θα φτιαχτεί. Έχετε λοιπόν μια τεράστια ευθύνη και ο Επίτροπος έχει τεράστια ευθύνη. τεράστια ευθύνη για σας να αλλάξετε την ατμόσφαιρα στο Συμβούλιο. Έχουμε ένα σημαντικό ραντεβού με την διάσκεψη Κορφής, με το Συμβούλιο να προχωρήσουμε και να εφαρμόσουμε το 1,5 βαθμό και ο Επίτροπος ξέρει πολύ καλά ότι αυτό σημαίνει την αλλαγή των στόχων μας για το 2020 γιατί ούτως ή άλλως τους έχουμε ξεπεράσει τους στόχους αλλά για το 2030 πρέπει να ε, καθαριστεί η αγορά του άνθρακα να γίνουν οικονομίες και να ενθαρρυνθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και έπειτα, ε, αν δεν το κάνετε αυτό, δεν θα κινηθεί το Συμβούλιο. Και ένα, μια τελευταία επιθυμία, κύριε Υπουργέ. Βλέπουμε μια μεγάλη ε, ε, κίνηση προς την έλλειψη επενδύσεων. Μήπως η Γαλλία μπορεί να αναλάβει μια μεγάλη πρωτοβουλία ε, με τις τράπεζες, με τους ιδιώτες. Πάρτε αυτή την πρωτοβουλία στο όνομα της Γαλλίας εν ώψη του Μαρακές. Έτσι θα συνεχιστεί αυτό το κίνημα. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο κύριος Αφρόντε παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ που είσαστε εδώ και για τη δουλειά που κάνατε στο Παρίσι. Όλοι εκτιμήσαμε την προσπάθειά σας. Η συμφωνία των πραγμάτων είναι συμβιβασμό, διότι υπήρχαν 195 χώρες γύρω από το τραπέζι, δεν μπορούσαν να γίνει διαφορετικά. Όπω κάθε συμβιβασμό έχει θετικά στοιχεία τα οποία επενθυμίστηκαν από εσά και του συναδέλφου, αλλά υπάρχουν και άλλα αρνητικά επί των οποίων θα πρέπει να στεστούμε. Και είναι απογοητευτικό ότι εξαφανίζεται η λέξη η απομάκρυνση τον θα πρέπει να σταματήσουμε να εκπέμπουμε. Βλέπουμε έναν ορισμό που είναι αμφίσιμο. Λέει να πετύχουμε ισορροπία μεταξύ των κομπών ανθρωπογενών και ε, τις εκπομπές αερίου του Δημοκηπίου. Μιλάμε για τεχνολογία αρνητικών εκπομπών. Αν τελικά θα μπορούσαν να εξισορροπήσουν τι θετικέ εκπομπέ, δεν ξέρω. Δημιουργήσαμε ένα άλοθη και είναι ένα άλοθη που προβλέπει τεχνολογίε προωθημένε και τεράστια χρήση των εδαφών. Στη, στην περίπτωση αυτή των συμφωνιών οι τεχνολογίε είναι επισήμω σημασία, αλλά τώρα είναι σε ένα πολύ πειραματικό στάδιο και πάρα πολύ δαπανηρό και δεν γνωρίζουμε θα λειτουργήσουν αυτέ τι τεχνολογίε στη στιγμή που δεν λειτουργούν και δεν ξέρω λειτουργούν παντού. Λοιπόν, θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η πραγματική δυνατότητα εφαρμογή όλων αυτών των τεχνολογιών με αρνητικέ εκπομπέ όσον αφορά τη μέγιστη κλίμακα εφαρμογή και ποια μέτρα παίρνουν οι κυβερνήσει για να διευκολύνουν αυτή τη δικασία. Ένα άλλο σημείο είναι η αγορά. Το σύστημα ETS, ανταλλαγή ρήπων, είναι ένα σύστημα κατά την άποψή μα δεν λειτουργεί. Δεν κατάφερε να τονώσει τι επενδύσει σε τεχνολογίε για να μειωθούν οι εκπομπέ και επ' αυτού έχουν γίνει κερδοσκοπίε και απάτε οικονομικέ. Θα πρέπει να υπάρχει παγκόσμια αγορά όπω λέει η Συμφωνία των Παρισίων και είναι κάτι μα μας ανησυχεί περισσότερο τις καθυστερήσει που θα δημιουργούσαν όσον αφορά την εφαρμογή άλλων πολιτικών που στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν μια πιο μεγάλη συνέπεια όπω τα κίνητρα για ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και τα μέτρα εξοικονόμηση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Και τέλο, θα πρέπει να κλείσουμε ένα κενό που υπάρχει μεταξύ αντίληψη πραγματικότητα και τη πραγματικότητα. Διαφορετικά θα εφαρμόσουμε αλλαγέ πάρα πολύ αργά. Με αργού ρυθμού. Το άρθρο 12 τη συμφωνία είναι καλό και το καλωσορίζουμε. Θα πρέπει να εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα και θα πρέπει να στέλνουμε ακριβή μηνύματα και αναλογικά προ τα προβλήματα. Θα πρέπει να γίνουν αυτά τώρα και θα πρέπει να απευθύνονται προ του πολίτε και την τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι και σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να γίνει προσπάθεια, θα πρέπει να γίνει κατανοητή κατανοητό ότι αυτό που παίζετε τώρα ε, δεν μπορούμε να παίζουμε άλλο, δεν υπάρχει χρόνο. Σα ευχαριστούμε κυρία Φρόντε. Στη συνέχεια ο κύριο Στούγκερ παρακαλώ. Μάλιστα πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρθηκε στην Γερμανία κάτι το οποίο γνώριζαν όλοι. Τότε δηλαδή ο τύπος βρίσκεται στα χέρια της ε, ελίτ που έχει την εξουσία όταν γράφεται κάτι για τους πρόσφυγες για παράδειγμα ή όταν πρόκειται για, για το κλίμα βλέπουμε ότι το πιο δυσμενές σενάριο παρουσιάζεται. Αν συνδέσει κανείς αυτά τα δύο θέματα καταλήγουμε με τους πρόσφυγες και τις κλιματικές αλλαγές ε, στον όρο κλιματικοί πρόσφυγες, ε, κλιματολογικοί πρόσφυγες. Ε, εδώ πρόκειται για παράδειγμα ένα ολόκληρο κινητήρα προπαγάνδας που παρουσιάζει και δίνει κάποιες λύσεις για όλα τα προβλήματα λέει που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ωστόσο, ο όρος και η προσέγγιση αυτών των κλιματολογικών προσφύγων είναι κάτι το οποίο μπορεί να ισχύει μόνο αν υπάρξει αυτή η υπερθέρμανση του πλανήτη. Ε, ε, και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι απογοητεύονται οι πολίτες και στρέφονται κατά των προσφύγων και αυτό είναι πολύ αρνητικό. Τώρα ο μη εγγεγραμμένος Μπαλτσό, κύριος Ευρωβουλευτής Μπαλτσό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Στις 15 Δεκεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε καταλεπτός ε, τα αποτελέσματα της ε, Συνόδου Κορυφής των Παρισίων, της διασκέψεως των Παρισίων. Γιατί πρέπει και πάλι να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Προφανώς, μάλλον, για να μπορέσει να ευχαριστήσει το Κοινοβούλιο τον Υπουργό κύριο Φαμπίους. Όλοι ευχαριστούν όλους. Πολύ ωραία όλα αυτά. Υπάρχουν όμως και κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν ακόμα απαντηθεί. Ποιο είναι το πραγματικό βάρος λοιπόν αυτών των υποσχέσεων που δόθηκαν και αναλήφθηκαν εκεί. Και τι θα συμβεί αν κερδίσει ένας ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος στις ε, προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το 2016 γνωρίζουμε ότι οι ρεπουμπλικανοί δεν συμμερίζονται τις ανησυχίες τις κλιματολογικές που έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Και τι θα συμβεί λοιπόν. Το πρωτόκολλο του Κιώτο δεν έχει ακόμα επικυρωθεί. Και ένα άλλο ερώτημα. Όταν και αν ε, υποστηρίζει σε θέματα ε, συναφή η Ευρωπαϊκή Ένωση τις αναπτυσσόμενες χώρες Ουγγαρία για παράδειγμα πώς θα μπορούσε από την Ουγγαρία να υποστηρίζεται όντας η δεύτερη πιο ισχυρή οικονομική χώρα. Υπάρχουν λοιπόν αναπάντητα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για τις παρεμβάσεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Τον λόγο θα λάβει τώρα για να ολοκληρωθεί η συζήτηση και πάλι ο Υπουργός κ. Φαμπίους παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Euh, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ εκείνους που μίλησαν και εκείνους που δεν πήραν το λόγο. Ήθελα να σας πω κύριε Πρόεδρε ότι έχοντας ακούσει αυτά που άκουσα είμαι έτοιμος να έρχομαι καθημερινά εδώ διότι ήταν ε, πάρα πολύ ευχάριστα. Στρωμένος ο δρόμος με τριαντάφυλλα για μένα σήμερα. Λοιπόν, μου κάνατε κομπλιμέντα και σε μένα και στον κύριο Κανιέτε. Όσον αφορά τη γαλλική διπλωματία, τα κομπλιμέντα δεν ξέρω αν ανταποκρίνονται στα όσα έγιναν. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε στο θέμα του 1,5 βαθμού, των 2 βαθμών, των φιλοδοξιών που θέσαμε. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο και το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος τη συμφωνία αυτή είναι το εξής δεν θα μπορούσαμε να μην συμφωνήσουμε διότι οι προηγούμενες διασκέψεις δεν είχαν δώσει και παράδειγμα τελείας ε, επιτυχίας. Ποιος ήταν ο βασικός κίνδυνος που εντόπισα. Να συμφωνήσουμε, αλλά να συμφωνήσουμε πάνω στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή όσον αφορά τις ε, φιλοδοξίες. Όμως, όταν είμαστε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν ρυθμίστηκα τα πάντα αλλά να πετύχουμε μια συμφωνία μεταξύ 195 χωρών χωρίς αντίρρηση, ε, διότι ήταν ελεύθερος να εκφραστεί ο κόσμος και πάνω σε ένα περιεχόμενο που είναι πολύ φιλόδοξο, περί αυτού πρόκειται, αυτό αποτελεί την επιτυχία των Παρισίων. Και εκεί μπαίνει η έννοια τώρα των βαθμών, του 1,5 των 2. Θα είδατε ότι η διατύπωση δεν είναι η ίδια για τους δύο βαθμούς και για τον 1,5 βαθμό. Οι δύο βαθμοί δεν ήταν εύκολο να επιτευχθούν. Αντικατέστησα τον πρόεδρο Ολάντα στους G20 και είχα πολύ μεγάλη δυσκολία να πετύχω το στόχο των δύο βαθμών. Τι έγινε όμως τελικά. Δημιουργήθηκε μια δυναμική στη διεθνή διάσκεψη που τελικά ευνοεί τον πλουραλισμό. Ακούστηκαν ισχυρέ απόψει από τα μικρά νησιά, από του προσώπου του που είπαν ότι δύο βαθμοί καλοί και άγιοι είπαν, αλλά αν δεν βάλετε 1,5 βαθμό και αν δεν λάβετε τα μέτρα για να πάμε προς 1,5 βαθμό, λέτε δηλαδή, υπονοείτε ότι εμείς δεν θα υπάρχουμε πλέον. Δεν είναι πλέον θέμα αν μπορούμε να ζήσουμε καλά ή όχι. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θα καλυφθούμε από το νερό. Δεν θα μπορούμε να υπάρχουμε. Και ήταν πολύ ισχυρό το επιχείρημα και που έπεισε χώρες που δεν ήταν αυθόρμητα υπέρ του 1,5 βαθμού θα εκφράσω και με χειρονομίες αυτό θέλω να πω. Σήμερα όταν αθρίζουμε όλα τα μέτρα είμαστε στους τρεις βαθμούς περίπου σαν στόχο, να είμαστε ειλικρινείς. Και μέσω της συμφωνίας των Παρισίων και της αποφάσεως που ακολούθησαν, αποφάσεων που ακολούθησαν με μακρόπνο ορίζοντα περνάμε με μια τροχιά από τρεις βαθμούς σε μια τροχιά δύο βαθμούς και μετά ένα μισή βαθμό. Μέσω συγκεκριμένων δράσεων και μέσω ενός σημείου που υπογραμμίσατε πολλοί από εσά, μέσω τεχνολογικών καινοτομιών και επενδύσεων σημαντικών. Στην αρχή δεν ήμουν ο ειδικό για αυτά τα θέματα, πρέπει να το ομολογήσω. Αλλά είμαι εργατικός και βυθίστηκα στο θέμα και μελέτησα και είμαι πεπισμένο ότι θα γίνουν τεχνολογικές αλλαγές σημαντικέ που θα καταστήσουν διαφορετική την ιεράρχηση των θεμάτων των ενεργειακών. Πολύ το υπογραμμίσατε αυτό. Ήδη σε κάποιες περιπτώσεις οι ανανεώσιμες πηγές ενεργείας είναι πολύ φθηνότερες όταν αθροίζουμε άμεσο και έμεσο κόστος από ότι οι ε, ρηπογόνες ενέργειες όπως ο άνθρακας. Και όλο και περισσότερο θα κινούμαστε προς τα εκεί. Έχουμε τη φιλοδοξία. Απ' τη μια και παγκόσμια εμβέλεια τη σύμφωνη από την άλλη που συμπλήρωναν η μία πτυχή την άλλη. Δεν ήταν αντιφατικέ. Και αυτή είναι η επιτυχία των Παρισίων και κάποιοι από εσά σωστά αναφερθήκατε στις ενέργειε και θαλάσσιες μεταφορές. Και εκεί θα τα πω, θα κοφτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και με πολλά άλλα μέρη ήθελαν να αναφέρουμε τις διεθνείς μεταφορές στη συμφωνία. Αλλά γνωρίζετε ποιος είναι ο μηχανισμός. Ο μηχανισμός της συνένεσης διαφάνει ότι αυτό το σημείο ε, αντιμετώπισε πολύ μεγάλη αντίδραση, να τα πούμε σωστά με το όνομά του, από ανεωδόμε οικονομίε και από τι χώρε του κόλπου. Άρα δεν ήταν δυνατόν να πετύχουμε συνένεση. Αυτό δεν δημιουργεί κανένα εμπόδιο, δηλαδή μπορούν οι διεθνείς, ε, οι διεθνείς οργανισμοί των αερομεταφορών, η ΚΑΟ και το IMO, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα και η Διεθνής Οργάνωση Θαλασσίων Μεταφορών. Όσοι έχουν καλή θέληση θα κινητοποιηθούν προς σωστή κατεύθυνση ο ΙΚΑΟ θέλει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 να φτάσει σε μια συμφωνία, σταθεροποιηθούν οι εκπομπές των αερομεταφορών ε, μετά το 2020 και να μειωθούν ενδεχομένως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπορώ να εκφράσω συνέστημα, θα πρέπει να ηγηθεί στο θέμα και να προωθήσει ανάντι διάφορες συνενέσεις όσον αφορά τις καλές μεταφορές. Ε, πρέπει να γίνουν σεβαστές οι συμφωνίες των Παρισίων και θα πρέπει να ανοίξουν οι διαπραγματεύσει στα πλαίσια του IMO και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ευνοήσει την αναγνώριση των εκπομπών του θαλασσίου τομέα, των τομέα των θαλασσίων μεταφορών και θα πρέπει να ενταχθεί στο παγκόσμιο σύστημα εκπομπών. Αλλά έχετε δίκιο. Επειδή έχουμε μεγάλε εκπομπέ από τον τομέα αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει φέτο να γίνουν σημαντικέ πρόοδοι όσον αφορά του δύο τομεί. Πολλοί από εσά σωστά αναφερθήκατε στο θέμα λίγο άνθρακα, πολλής άνθρακα, ανταγωνιστικότητα κλπ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι κεντρική σημασία. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Δηλαδή, και αντίθεση. Εκπομπέ αερίου του θερμοκηπίου από την άλλη πλευρά και από την άλλη χρειαζόμαστε να έχουμε και ανταγωνιστικότητα παράλληλα. Και χρειάζεται να έχουμε και απασχόληση. Χρειάζονται αλλαγέ, μεταμορφώσει, συνοδευτικά μέτρα κλπ. Αλλά είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι η ανταγωνιστικότητα όχι μόνο για τις χώρες όπως είναι οι δικές μας, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να παντρευτεί με μια πρόοδο προς τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Και εδώ ε, απαντώ και στο ερώτημα του κ. Ζαντό νομίζω που το έθεσε των, ε, των επενδύσεων. Ήδη είδατε ότι πέρα από τι επενδύσει του δημόσιου τομέα που είναι κάτι πολύ σημαντικό και στον δυτικό τομέα υπάρχει μια αλλαγή που λαμβάνει η χώρα. Τόσο το καλύτερο. Θα πρέπει να μπορέσουμε να επιταχύνουμε. Πιστεύω θα πρέπει οι, οι χώρες να μειώσουν σταδιακά τις επιδοτήσεις υπέρ των, ορεικτών των ε, καυσίμων. Αυτή η αρχή καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαΐου του 2013 και η Γαλλία είχε ζητήσει φιλόδοξο στόχο όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις για ε, τις μονάδες άνθρακα. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου είναι χαμηλές. Γνωρίζετε τα στοιχεία. Μιλάμε για 100 δις που θα πρέπει οι πλούσιες χώρες να διαθέσουμε για το κλίμα προς τις φτωχές χώρες. Αλλά τα ποσά που αφιερώνονται από τις επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα ε, ξεπερνάνε τα 500 δις. Άρα έχουμε περιθώρια. Μετά για να απαντήσω στον κύριο Ζαντού θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους φορείς του ιδιωτικού τομέα να μην επενδύουν, να μειώσουν τις επενδύσεις στον τομέα που χρησιμοποιεί πολύ άνθρακα. Και από την COP21 είδαμε ότι δημιουργήθηκε μια κίνηση. Το πρώτο, το Νορβηγικό Ταμείο έδωσε ενδείξει να μειωθούν οι επενδύσει και ο διευθυντή τη Βρετανική Κεντρική Τράπεζα είπε ότι η επόμενη φούσκα οικονομική θα μπορούσε να δημιουργηθεί στον τομέα αυτό του άνθρακα διότι αυτό ο τομέα σίγουρα θα αντιμετωπίσει δυσκολίε ενώ επενδύσει τεράστιε ε, γίνονται εκεί σε αυτό το τομέα του άνθρακα. Τώρα όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα μπορούμε να ζητήσουμε από τις κεντρικές τράπεζες και τους φορείς βαθμολόγησης να λάβουν υπόψη συστηματικά τον κίνδυνο που δημιουργείται όσον αφορά το κλίμα και είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των ιχνο, του ίχνους άνθρακα. Ε, και αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Παράλληλα με αυτή την τάση μειώση των επενδύσεων θα πρέπει να γίνει προσπάθεια προς τις επενδύσεις στις ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μέσα το σχέδιο Juncker, τα διευθυντικά ταμεία, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που θα πρέπει να κινητοποιηθούν. Έχετε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει τον Μάρτιο και από αυτή την ευκαιρία πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε μια αξιολόγηση εφαρμογή και υλοποίηση συμφωνία των Παρισίων. Είναι διάφορε κατευθύνσει προ τι οποίε μπορούμε να κατευθυνθούμε. Δεν θα μακρηγορήσω. Τελευταίο σημείο αφορά τα κομπλιμέντα που μου που απευθύνατε όσον αφορά τη σύνεση την οποία κινηθήκαμε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρόλος του όπου του κυρίου Κανιέτε, ο ρόλος της Προεδρίας του Λουξεμβούργου είναι κάτι που εγκρίνουμε ανεπιφύλακτα. Αντίθετα τώρα, όσον αφορά τη γαλλική διπλωματία, ακόμα και αν αυτή μέσω εμού ε, ερυθριά ακούγοντά σα, διότι είμαστε πολύ μετριόφρονες, αυτό είναι τη πάση γνωστό, Σκεφτόμουν όμως ε, ρόλος σας και ρόλος μου ποιος ήταν να ευνοήσουμε, να βοηθήσουμε ούτω ώστε να επιδευτεί μια αξιοσημείωτη ευθυγράμμιση στον πλανήτη. Το 2015 ήταν ο πιο θερμός χρόνος για τον πλανήτη με πολύ σημαντικές καταστροφές και η κοινή γνώμη ευαισθητοποιήθηκε. Αυτή η καταστροφική λοιπόν κατάσταση έχει και μια καλή πλευρά, αν μπορώ να το πω έτσι. Έγινε προφανέστερη ακόμα η ανάγκη ύπαρξη συμφωνίας. Και αυτό ευνόησε την ευαισθητοποίηση, τη συνειδητοποίηση. Ο πρώτος πλανήτης, ο δικός μας ο πλανήτης λοιπόν, μας οδήγησε σε αυτή την ευθυγράμμιση. Ο πρώτος πλανήτης λοιπόν. Δεύτερο δεύτερος είναι ο επιστημονικός πλανήτης. Από τι φόρο τιμής λοιπόν στις ε, αξιέπαινες εργασίες των επιστημόνων που έδειξαν αδιαφυσβήτητα ότι ε, αυξάνεται η θερμοκρασία και έγινε προσμέτρηση των συνεπειών. Όταν κάναμε συνεδριάσεις πριν, η μισή συνεδρίαση εξετάσαμε κατά πόσο υπήρχε αναστάτωση του κλίματος και στο δεύτερο τμήμα της συνεδριάσεως ε, προσπαθούσαμε να δούμε ένα ανθρωπογενή αποτελέσμα. Τώρα πια δεν λέω ότι έχει ε, λήξει αυτή η συζήτηση, αλλά έχει μειωθεί σημαντικά αυτή η αμφισβήτηση. Και χάρη στη δουλειά των επιστημόνων έγινε αυτό. Και αυτό ο επιστημονικό πλανήτη, αν θέλετε να βοήθησε μετά, τρίτο πλανήτη που υπάρχει, θα είναι ο πολιτικοκοινωνικό πλανήτη. Ε, υπήρχαν ε, χώρε που εξέπεμπαν πάρα πολύ μεγάλε ποσότητε αερίων θερμοκηπίου. Η Κίνα, πρώτη εκπομπέ, που για λόγου προφανεί, πρακτικού, οικονομικού, κοινωνικού, και επιχειρηματικούς έπαιξε ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό. Ο πρόεδρος Ομπάμα ανέλαβε δεσμεύσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια και άλλες χώρες. Επέτρεψε τελικά η κατάσταση να υπάρξει μια μεγάλη μετακίνηση των οικονομικών κύκλων. Οι κοινότητες δεσμεύτηκαν, οι περιφέρειες δεσμεύτηκαν, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεσμεύτηκαν οι μεγάλοι θρησκευτικοί ηγέτες και τα κύματα, ε, κύκλοι κινητοποιήθηκαν. Και αυτό είναι ο πλανήτης, ο κοινωνικοπολιτικός που ανέφερα, που κινητοποιήθηκε. Και στη διάσκεψη των Παρισίων είχαμε διαφορετική προσέγγιση σε σύγκριση με τη διάσκεψη της Κοπενχάγης. Τέτος πλανήτης είναι ο διπλωματικός, θα έλεγα. Καθήκον μας ποιο ήταν, μαζί με όλες τις χώρες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Θέλαμε να ευνοήσουμε τη σύγκληση και όλα αυτά να μεταφραστούν σε μια διεθνή συμφωνία με τα 29 άρθρα και τα 140 σημεία αποφάσεων. Και διερωτώ με συχνά τι πιάνει η δουλειά που έκανε διπλωμάτες κλπ. Αστεζόμενος λέγω ότι δεν καταλάβαινα απόλυτα τους λόγους της επιτυχίας, αλλά προτιμώ να μην καταλαβαίνω τους λόγους της επιτυχίας παρά να έχω εξηγήσει λαμπρές για μια αποτυχία. Από τη στιγμή το λέω αυτό μεν, αλλά ουσιαστικά όταν επενεξετάζω τη δουλειά που κάναμε είδα ότι ήταν σαν να κινηθήκαμε σαν γλύπτες. Παίρνει ο γλύπτης ε, το πυλό, ένα κομμάτι ε, πύλου. Παίρνει τα βασικά κομμάτια, ας πάμε τα κομμάτια ποια ήταν η Κίνα, η ΙΠΑ, η Ευρώπη εδώ, η Ινδία. Και έπρεπε λοιπόν να τα συναθρήσουμε τα κομμάτια και να δώσουμε κάποια μορφή στα κομμάτια. Και μετά τα πιο μικρά κομμάτια που χρειάζονται και αυτά τα μικρά κομματάκια διότι δεν υπάρχει συνένεση, δεν υπάρχει συμφωνία χωρίς συνένεση. Και έπρεπε να δώσω μια μορφή σε όλα αυτά χωρίς να χάσουμε κανένα από τα κομμάτια. Αυτή ήταν ε, η δουλειά που κάναμε σε ένα πνεύμα διαφανείας και εμπιστοσύνης, κάτι που υπογραμμίστηκε και στο τέλος αυτό το θέαμα ε, θα δώσω ε, ένα μικρό σφυράκι στον κύριο Σούλτς που είναι και το πιο περίφημο, το πιο διάσημο σφυράκι που χρησιμοποιήθηκε και στο τέλος ε, όλοι αγκαλιαστήκανε στις διεθνούς διάσκεψεις. Δηλαδή, είχαμε την εντύπωση σε ένα πολύ σκληρό, επικίνδυνο, περίπλοκο και αβέβαιο κόσμο, για πρώτη φορά, χάρη στην προσπάθεια όλων, ε, έγινε κάτι που πραγματικά που επέτρεπε όχι μόνο στην παρούσα γενιά, αλλά και στις μελλοντικές γενιές να ζήσουν καλύτερα. Και όπως ε, υπογραμμίστηκε, προφανώς είναι περιστάσεις που δεν αντιμετωπίζουμε πάντα πολιτικό στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ όλους που το καταστήσατε αυτό εφικτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με αυτή την